Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν ε, ε, στο Κοινοβούλιο για έγκριση. Αν δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις, οι προτάσεις ψηφίσματος που εγκρίθηκαν σήμερα θα διαβαστούν αρμοδίως. Και εδώ μπορώ να κηρύξω τη λήξη των εργασιών της Ολομέλης αυτής.